δραστηριότητες για το μέλλον. Στις αρχές του 2014, όπως σας είπα, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 12 μεσημέρι. Τώρα, στην ημερήσια διάταξη έχουμε την κοινή συζήτηση για τα οχήματα, έχουμε την έκθεση Vandenkamp ε, για την αγορά δίκυκλων ή τρικυκλών χυμάτων και τετράκυκλων, έγκριση και αποπτία της αγοράς και έχουμε και την έκθεση Παντσέρη για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων για τέσσερα λεπτά. Το λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Vandenkamp. Παρακαλώ. Mevrouw de voorzitter, eh, dank Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα κύριε Ταγιάννη, καλησπέρα στους βοηθούς σας. Κυρία Πρόεδρε, εδώ έχουμε ένα τεχνικό φάκελο, ο οποίος εκκρεμεί εδώ και καιρό. Αλλά είναι πολύ σημαντικός για την εσωτερική αγορά. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνικές προδιαγραφές στα δίκυκλα, αλλά πρόκειται και για την εποπτεία τους. Για να αρχίσω από το πρώτο θέμα, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τελευταία δύο χρόνια συζητήσαμε πέντε σημεία που δημιούργησαν μετά τον κανονισμό. Πρόκειται για την κατηγοριοποίηση των οχημάτων και πρέπει αυτό να το διευκρινίσουμε. Συζήτησα με τον συνάδελφο Πανσέρη για τα επαγγελματικά οχήματα, μετά μιλήσαμε για τα συστήματα πέδησης, ε, το ABS και το CBS, στα δίκυκλα οχήματα. Αυτά τα συστήματα πέδησης πρέπει να γίνουν ασφαλέστερα. Σε ό,τι αφορά τα μικρά σκούτερ πρέπει να γίνει μια μελέτη αν εκεί είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα ή όχι. Επίσης είδαμε το θέμα των εκπομπών των οχημάτων γιατί το, γιατί είναι υψηλές οι εκπομπές τους. Επίσης είδαμε και τα τεστ βιωσιμότητας, γιατί ένα μικρό ε, δίκυκλο πρέπει να είναι ε, εξίσου ασφαλές στη διάρκεια των ετών, όπως και η φανή του. Επίσης, ε, είναι σημαντικό, κυρία Πρόεδρε, τα ε, δίκυκλα που έχουν άδεια στην Κίνα και την Ινδία να μην έρχονται στην Ευρώπη και όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά για την ποιοτική ασφάλεια των πολιτών μας. Πριν συνεχίσω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετασχόντες στη συζήτηση και τη Δανέζικη Προεδρία που ασχολήθηκε πολύ με το θέμα αυτό. Επίσης ευχαριστώ Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ορισμένα ερωτήματα προς τον Επίτροπο για τις διαπραγματεύσεις, για τις ε, εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Συμφωνήσαμε να έχει χρόνο η οικονομία για να εφαρμόσει τον νέο κανονισμό. Αλλά αν διαρκέσουν πολλοί διαδικασίε των εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξεων, τότε δεν θα μείνει πολύ καιρό για την οικονομία, για τον κλάδο. Θα ήθελα να με διαβεβαιώσει ο Επίτροπο ότι η Κομισιόν θα επιτελέσει πρόοδο με τι δύο αυτέ πράξει, εκτελεστικέ και κατεξουσιοδότηση. Δεύτερον, οι απαιτήσει εκπομπών Euro 5 κατηγορία το 2016. Η Κομισιόν πρέπει να διεξαγάγει μελέτη εδώ. Δεν ε, πρέπει να δούμε μόνο τους ρήπους αλλά και το κόστος και πάλι πρόκειται για το lead time. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει κάποια ασάφεια σε σχέση με τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή αυτής της οδηγίας αλλά πάνε στην οδηγία για τα μηχανήματα. 25 ε, χιλιόμετρα την ώρα. Ε, ε, αυτά θα πρέπει να καλυφθούν γιατί μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα. Ε, ενδεχομένως μπορεί αργότερα να συμπεριληφθούν. Είχαμε επαφές και με τη μητρική κατασκευαστική εταιρεία που ήταν πολύ επικριτική. Ε, καλό είναι για την δημοκρατία αν ε, μας επικρίνει η μητρική αγγλική κατασκευάστρια εταιρεία. Ε, δεν λέω, θα πρέπει να γίνουν αλλαγές αλλά όχι προς επιταχύρω. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Εγγλέζοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τέσσερα λεπτά στον κύριο Παντσέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νομοθετική διαδρομή ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2010. Ήταν ε, μια πολιτική και τεχνική δουλειά αρκετά δύσκολη που διήρκησε δύο χρόνια και ασχολήθηκαν με αυτή τρεις προεδρίες του Συμβουλίου. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συμμετείχαν, τους συναδέλφους και συζητές, τη γραμματεία, τις πολιτικές ομάδες, ε, τους συνεργάτες των βουλευτών και φυσικά την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Για το τελικό κείμενο υπάρχει μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση, αυτό το θεωρώ κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός ο κανονισμός έχει στόχο να δημιουργήσει μια σειρά εναιμονισμένων κανόνων ε, για την κατασκευή γεωργικών και δασικών οχημάτων προκειμένου να εγγυθούμε την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εγγυθούμε την εφαρμογή πολλών και σημαντικών κριτηρίων που βελτιώνουν ε, την λειτουργία της, ε, την ασφάλεια της χρήσης ε, αλλά και την ασφάλεια στους δρόμους όπως και τα περιβαλλοντικά πρότυπα έτσι ε, το ότι έχουμε στα άρθρα 6 και 7 νέε απαιτήσει επαγγελματικού χαρακτήρα αλλά και λειτουργικού χαρακτήρα μπορεί να θεωρηθεί πραγματική επιτυχία για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατόρθωσε να καλύψει αυτού του κινδύνου που σήμερα θίγουν ε, πάρα πολλού ε, χρήστε πολύ συχνά με κάποιε θανατηφόρε συνέπειε κατά τα λοιπά. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε το θέμα τη ασφάλεια και τη υγεία των εργαζομένων και γι' αυτό έχουμε προβλέψει κάποιες διατάξεις σχετικά με την εποπτεία της αγοράς οχημάτων, συστημάτων ε, και εξαρτημάτων για να εγγυηθούμε ότι όλες οι διατάξεις που προβλέπονται θα, είναι, θα, θα σε σωστή εφαρμογή. Ο κανονισμός τέλος συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, του κλάδου, γιατί απλοποιεί τη σημερινή νομοθεσία για την έγκριση τύπου, αυξάνει τη διαφάνεια και μειώνει το διοικητικό ε, ανακαλούνται 24 βασικές οδηγίες και περίπου 5 οδηγίες τροποποίησης σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσει και όλα αυτά τα αντικαθιστάνε και μόνος κανονισμός. Αυτές οι σημαντικές πτυχές ε, είναι σημαντικέ πτυχέ γιατί μέσω του κανονισμού θέλουμε να πετύχουμε και κάποιου άλλου στόχου πέρα από την οικοδόμηση μια ρυθμισμένη εσωτερική αγορά και τη υλοποίηση ενό συστήματο ισορροπημένου και διαφανού. Πέραν αυτού συνεισφέρουμε στην ενίσχυση του κλάδου και τελικά δημιουργούμε τις συνθήκες για να διευρυθεί η παραγωγική βάση και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Έτσι λοιπόν το έργο που έχει υλοποιηθεί είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ιδιαίτερα καρποφόρο οι δεσμεύσεις, που, οι συμβιβασμοί που επιτεύχθησαν από όλε τις πολιτικές ομάδες μας έδειξαν ότι υπήρξε το σωστό πνεύμα συνεργασίας και υπήρξε βούληση τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξει σε ένα κανονισμό στο οποίο όλοι συμφωνούν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Σταγιάννη. Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι πάρα πολύ που παρευρίσκομαι εδώ κυρίως ε, γιατί ολοκληρώνεται μια μακρά και δύσκολη διαδρομή νομοθετική για την έγκριση δύο νομοθετικών κειμένων, πολύ σημαντικών, από τεχνική σκοπιά, που χρησιμεύουν και στην ε, ελάφρυνση της σημερινής νομοθεσίας ε, και σε ό,τι αφορά την έγκριση τύπου για τα δασικά και αργικά οχήματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί είχα ε, δεσμευτεί κατά την ακρόασή μου ε, ως υποψήφιος επίτροπος και χαίρομαι πάρα πολύ που η δέσμευση που είχα λάβει την τήρησα. Και μάλιστα χαίρομαι που έχουμε και την συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις μακρές διαπραγματεύσεις, όπως είπε και ο κύριος Πεντσέρη, είχαμε θετικά αποτελέσματα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους δύο εισηγητές αλλά και τους και εισηγητές. Τα συμβιβαστικά κείμενα αποτελούν αποτέλεσμα μια σειρά συζητήσεων επικοδομητικών και με την Επιτροπή και το Συμβούλιο που διήρκησαν σχεδόν δύο έτη γιατί όπως είπαμε πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο ζήτημα από τεχνική σκοπιά. Θέλω να υπογραμμίσω ότι οι νέοι οικονομισμοί θα βελτιώσουν σημαντικά ε, την ασφάλεια και το σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον θα ωφελήσουν τους πολίτες ε, και την κοινωνία και επίσης έχουμε και αρκετό χρόνο για να επιτρέψουμε στον κλάδο να προσαρμόσει την παραγωγή στις νέες απαιτήσει. Ε, Έχουμε κάποιες απλουστεύσεις στο νομοθετικό κείμενο που θα επιτρέψουν και τη μείωση του κόστους. Έτσι λοιπόν κατορθώσαμε να έχουμε μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων. Η οθέτηση αυτών των δύο νομοθετημάτων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα μπρος για την απλούστευση και για την καλύτερη νομοθεσία και για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς όπως ε, υπογράμμισαν και δύο οι δύο κανονισμοί αποτελούν, μάλλον αντικαθιστούν 40 οδηγίες ε, και σε αυτές έχουμε μία σειρά κατεξουσιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών πράξεων. Εγώ σημείωσα τόσο είπε ο κ. Βαντεκάμπ, επομένως θα ακολουθήσουμε και την πτυχή που υπογράμμισε ο εισηγητής. Επίσης προβλέπεται να βελτιωθεί η συνοχή μεταξύ δύο καθεστώτων έγκρισης τύπου. Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία των δύο κειμένων. Καταρχήν, έχουν εισαχθεί κάποιε διτάξει για την πρόσβαση στι πληροφορίε ε, σχετικά με τι επισκευέ και τη συντήρηση για να εγγυθούμε ότι ενημερώνονται σωστά οι καταναλωτέ. Κατόπιν, έχουμε απαιτήσει εποπτεία τη αγορά. Τρίτον, έχει εισαχθεί μία κατηγοριοποίηση των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων. Κυρίω έχουμε ε, τα επαγγελματικά οχήματα παντού εδάφου και τα οχήματα αναψυχή εκτό δρόμου που μπορούν να μπουν στη κατηγοριοποίηση και των διοκανονισμών αν σέβονται του ορισμού και τα τεχνικά στοιχεία, τι τεχνικέ απαιτήσει. Επίση, βελτιώθηκε η προστασία του περιβάλλοντο και η ασφάλεια των οχημάτων αυτών. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειε για τι μεμονωμένε προτάσει, γιατί έχει γίνει αυτό με σαφήνεια από του συζητητέ μα. μόνο ορισμένα σημεία ανέφερα τα οποία συμφωνήσαμε με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επαναλαμβάνω επειδή μου επιτρέψετε να τηρήσω μια δέσμευση που είχα λάβει ενώπιον σας και ενώπιον των πολιτών. Και πιστεύω ότι αυτό ωφελεί τα θεσμικά όργανα κάποια στιγμή που πολλέ φορέ υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντί μα. Ε, το να εργαζόμαστε ορθά και να τηρούμε τι υποσχέσει μα ε, σημαίνει ότι απαντούμε συγκεκριμένα στα μηνύματα που μα έρχονται από πολλά μέρη τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Τώρα ε, Τζίλα για δύο λεπτά από την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε να συγχαρώ τον εισηγητή Βιμ Βαντε Κάμπ για την συμφωνία στο Κοινοβούλιο. Στην Επιτροπή Μεταφορών εξετάσαμε από την άποψη της ε, οδικής ασφάλειας το θέμα, γιατί τα δίκυκλα είναι το 60% των ε, τροχαίων θανάτων στην Ένωση. Χαιρετίζουμε επίσης το γεγονός ότι το κείμενο που συμφωνήθηκε αντιμετωπίζει ε, άριστα τα θέματα των προδιαγραφών ασφαλείας όλων των δίκυκλων και προβλέπονται και τεχνικές, ε, προ... Ε, τεχνικές προϋποθέσεις για οδική ασφάλεια. Αυτή ήταν μία από τις προτάσεις ε, της Επιτροπής Μεταφορών να γίνει μετακανονισμός. επίσης, τα οχήματα ε, που κυκλοφορούν σε δημόσια οδικά δίκτυα πρέπει να καλύπτουν όλα αυτά τα συστήματα. Η Επιτροπή ε, Μεταφορών θεωρεί για τα δίκυκλα ότι ε, η επίτευξη της βέλτιστης ασφάλειας είναι πρώτη προτεραιότητα. Η μελέτη επιπτώσεων μπορεί να ε, δείξει και τα, την απόδοση των συστημάτων πέδησης ε, και αυτό θα πρέπει να το καλύπτει ο κανονισμός. Τέλος, στηρίζω την πρόταση, τη λύση που βρέθηκε για το, ε, τις καινούργιες κατηγορίες ε, ε οχημάτων Euro σε αυτή την κατηγορία. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχουν εκπροσωπεί των πολιτικών ομάδων. Γκάλ Πέλτ για το ΕΛΚ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ τον κύριο Βάντε Κάμπ για την έκθεση. Έχω την αίσθηση ότι η πρόταση αυτή πραγματικά ε, στρέφει την προσοχή στον τομέα, αυτό είναι σημαντικό, στρέφει την προσοχή στο γεγονός ότι κατά την κατασκευή οχημάτων πρέπει να συντρέχουν σημαντικές προϋποθέσεις. Πρέπει να προσέξουμε στη ρύθμιση αυτή ο τομέας των κατηγοριών 2 και 3 να ε, τηρεί τις ε, προδιαγραφές του 90% της ευρωπαϊκής παραγωγής ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος επιχειρήσεων. Αυτό έχει να κάνει και με τις θέσεις εργασίας. Το 10% είναι μικρές επιχειρήσεις σε διάφορα κράτη-μέλη. Υποθέτω λοιπόν ότι οι ε, λήψεις μέχρι τώρα ε, οφείλονταν και σε ελλειπείς ε, νομοθεσίες αλλά και πρότυπα και προδιαγραφές που καθορίστηκαν το 2006. Η Κομισιόν προτείνει και άλλες βελτιώσεις και έτσι σταδιακά εισάγει καινούργια μέτρα. προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τη βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων. Επίσης πρόκειται και για την τήρηση των στόχων ε, του 2012, από το 2012. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι ασχοληθήκαμε με το κείμενο αυτό για να επιτευχθούν οι σωστοί στόχοι. Για τη ρύθμιση τώρα των λειτουργίας εσωτερικής αγοράς είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν σωστά οι τεχνικές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες σε ό,τι αφορά την επισκευή των οχημάτων. Θα πρέπει να είναι σωστός ο ανταγωνισμός και να υπάρχουν πληροφορίες σε σχέση με την λειτουργία των οχημάτων και τις επιδόσεις τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σημαντικές και τα στοχευμένα μέτρα που πρέπει να αποφασίσουμε είναι επίσης σημαντικά. Αυτά θα πρέπει να είναι σωστά και να έχουν σωστή επίπτωση για τις ε, μικρομε... να έχουν τις σωστές ε, επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχει πολλά σημαντικά και καλά και θετικά σημεία η έκθεση και τα μέτρα εποπτείας της αγοράς είναι και αυτά σημαντικά, όπως και η, ε, δημιουργία ενός ε, συστήματος εδώ. Η... Τα οχήματα που έγκρισης τύπου και μη έγκρισης τύπου, αυτή η διαφοροποίηση είναι πολύ σημαντική. Παράλληλα καλύπτεται εδώ και ο τεχνικός έλεγχος. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι στην έγκριση των ε, τύπων οχημάτων μπορούμε να επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ άλλη μια φορά τον εισηγητή και έχω τη γνώμη ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα πράγματα ε, παρά μόνο να κινηθούμε προς το συμφέρον της καλύτερης δυνατής εφαρμογής στην πράξη των μέτρων αυτών και των διατάξεων που θεσμοθετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ε, συνάδελφος Βέστβαλ, ε, για 4,5 λεπτά. Κυρία Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε ότι αυτό που πήρε πολύ χρόνο, στο τέλος ε, κατέληξε καλά. Η έκθεση αυτή έγινε πάρα πολύ καλή. Οι εργασίες διήρκεσαν περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε και ελπίζαμε όλοι. Και ε, υπήρχαν ε, πολλά, πολλές, σε πολλά σημεία ακολουθήσαμε λάθος πορεία. Όμως τώρα θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Βάντερ Κάμπ για την εξαιρετική συνεργασία. Μαζί στις διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη επιτύχαμε πολλά πράγματα. Ως εισηγήτρια για την ομάδα μου, ε, η σύστασή μου είναι να ψηφίσουμε υπέρ της έκθεσης, παρόλο που θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ καλύτερη. Και όταν λέω καλύτερη, εννοώ αγαπητοί συνάδελφοι, ε, να επιτύχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Για μας τους ε, σοσιαλδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτησες, ε, ευθύ εξ αρχής η ασφάλεια των οχημάτων και φυσικά έτσι και η ασφάλεια των οδηγών ήταν πάντοτε πρώτη προτεραιότητα. Ιδιαίτερα η ασφάλεια των δικύκλων μοτοσυκλετών. Ο αριθμός των ατυχημάτων ε, εδώ και χρόνια παραμένει σε, στα ίδια υψηλά επίπεδα. Ε, όμως στην Ευρώπη μειώνεται ο αριθμός των θανάτων από τροχέα ε, γενικότερα. Μόνο στα δίκυκλα όχι. Η μείωση των ε, θανάτων μοτοσυκλετιστών είναι για μας ένα θέμα πολύ σημαντικό. Λιγότεροι νεκροί στους δρόμους της Ευρώπης. Ήταν και είναι ο στόχος μου. Κάθε θάνατος, κάθε νεκρός είναι ένας πάρα πολύ. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να ωφελεί την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να τύχει ε, πολύ σημαντικής επεξεργασίας. Ε, αποτελεσματικά συστήματα πέδησης ε, ε, αντιεμπλοκής. Είναι πολύ σημαντικό. η σχέση ωφέλειας πρέπει επίσης να είναι πολύ σημαντική. Τα συστήματα αυτά δεν είναι αλήθεια ότι είναι πολύ ακριβά εμείς ε, πετύχαμε από το 2016 όλα τα καινούρια και από το 2017 όλα τα υφιστάμενα δίκυκλα ε, ε, πάνω από 250 κυβικά θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται από, με συστήματα πέδησης αντιεμπλοκής ABS από τον κατασκευαστή. στα ε, δίκυκλα ε, μπορέσαμε να το πετύχουμε αυτό. Ή ε, απέδηση αντιμπλοκής ή συνδυασμένα συστήματα απέδησης. δεν επιτύχαμε παντού βελτιώσεις σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα κάτι περισσότερο. Η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, για να το διατυπώσω προσεκτικά, αποδείχθηκαν πολύ δυσκίνητα. Καταφέραμε όμως ε, το 2019 η Κομισιόν να υποβάλει μια έκθεση. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να ε, έχει ε, στοιχεία για τα τροχέα από τα κράτη-μέλη και θα πρέπει να εξετάσει την εγκατάσταση συστημάτων πέρυσις αντιεμπλοκής τα συστήματα ABS. Στη βάση αυτής της έκθεσης η Κομισιόν θα σκεφτεί μετά να ενσωματώσει το σύστημα ABS υποχρεωτικά στα δίκτυα αυτά βλέπουμε ότι το, το θέμα αυτό παραμένει πάρα πολύ ζωντανό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν από το 2019 αυτό το υποχρεωτικό κενό στην νομοθεσία να το κλείσουμε. Είμαι βέβαιη ότι τα στοιχεία που θα συλλέξουμε θα με δικαιώσουν. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή είναι μια καλή ημέρα για τους τις οδηγούς δικύκλων στην Ευρώπη και ότι στο μέλλον θα μειωθεί και ο αριθμός των τροχαίων ε, ατυχημάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους φιλελεύθερους. Μάντερς για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, ειδικότερα τους κυρίους Βαντενκάμπ και Μπεντσέρη για τις εισηγήσεις τους με σκοπό τη βελτίωση της αγοράς, ε, τη δημιουργία καλύτερου περιβάλλοντος με μεγαλύτερη σαφήνεια για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, χαμηλότερο κόστος διοικητικό και λιγότερους κανόνες. Και ως ε, φιλελεύθερος αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το θέμα αυτό αποδείχθηκε ιδιαίτερα τεχνικό και εγώ αισθάνομαι λιγάκι σαν τεχνοκράτης και τα πράγματα τόσο δύσκολα κάποια στιγμή, είχαμε τόσες πολλές τροπολογίες που ένιωθα σαν τεχνικός και όχι πλέον σαν πολιτικός. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερο, περισσότερο πολιτικό στοιχείο σε αυτή την υπόθεση. Στο μέλλον θέλουμε να μπορούν να αλλάχθουν οι μπαταρίες σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων. Θέλουμε να προωθήσουμε την καινοτομία ή θέλουμε να παγώσουμε τα πάντα στα πλαίσια της ε, σε τύπου. Πώς θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια. Πώς μπορούμε <clears throat> να καταπολεμήσουμε τα κακά προϊόντα ή τα ερζάτς προϊόντα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Βαντεκάμπ. Θέλουμε να γράφουμε Made in Europe ή όχι πάνω στο όχημα. Μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η χώρα παραγωγής ο καταναλωτής. Πώς θα αποφύγουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, τα ε, τρακτέρ, τα γεωργικά μηχανήματα, μέρη μουλκούμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με, η έγκριση τύπου γίνεται πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με τα φορτηγά. Η ασφάλεια του οχήματο βεβαίω εξαρτάται από τη συμπεριφορά του οδηγού. Και εγώ θα ήθελα να καθορίσουμε ελάχιστου ευρωπαϊκού κανόνε που θα ισχύουν παντού στην Ευρώπη και θα αφορούν του οδηγού. Και επίση πρέπει να γίνεται τακτική ενημέρωση, μια, ε, διότι παίρνει κανεί την άδεια οδήγηση το δίπλωμα οδήγηση όταν είναι νέος, οι τεχνικέ αλλάζουν, οι συνθήκες κυκλοφορίας αλλάζουν και δεν είναι έτοιμοι οι οδηγοί σε πάρα πολλέ περιπτώσεις να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες συνθήκες. Θα ψηφίσουμε υπέρ, αλλά θα ήθελα να υπάρχει πιο έντονο ε, πολιτικό στοιχείο σε εκθέσεις σαν και αυτή, με μεγαλύτερη, με ε, μεγαλύτερη εστίαση σε αυτά που επιθυμούν οι καταναλωτέ. Ε, σας ευχαριστώ όλους και είμαι βέβαιος ότι ότι αύριο θα υπάρξει μεγάλη πλειοψηφία που θα ψηφίσει υπέρ αυτών των δύο ε, εκθέσεων. Ευχαριστώ. Ως πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, ήμουν σκιώδης και σε αυτούς τους δύο φακέλους και ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής ε, και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο ε, που ασχολήθηκαν με τόσο δύσκολα θέματα και ξέρω ότι ο κύριος Μπάντερς θέλει να τα παρουσιάσει πιο συναρπαστικά από πολιτική σκοπιά αλλά πρόκειται για πραγματικά σημαντικούς φακέλους και για τους δύο κλάδους και θα θέσουν το μοντέλο για ένα σύστημα έγκρισης τύπου πιο απλοποιημένο. Στην περίπτωση των μοτοσυκλετών νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι ε, συμβάλαμε στο να έχουν καλύτερες ε, επιδόσεις ε, ασφάλειας και περιβαλλοντικές ε, επιδόσεις οι μοτοσυκλέτες και τα οχήματα αυτά θα γίνουν πιο δημοφιλή στο μέλλον, θα συνεισφέρουν στο να έχουμε μεταφορές χαμηλών εκπομπών και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντερκάπ ιδίω γιατί διασφάλισε ότι στα σταδιακή περίοδος ε, το phasing in ε, θα ε, ήταν ουσιαστικά μία καλή περίοδος και θα είχαμε μεθόδους αποτελεσμα κόστος αποτελέσματος. Ε, τώρα για τα τρακτέρ, ε, εκεί έχουμε συμπεριλάβει και τα γεωργικά και δασικά οχήματα. Έχουμε μια πολύπλοκη σειρά κανόνων και κανονισμών εκεί, αλλά τώρα έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα έγκρισης τύπου που θα βοηθήσει τους κατασκευαστές και υπάρχουν και πολύ μικρά κατασκευαστές σε αυτό το τομέα να παρουσιάσουν προϊόντα για έγκριση τύπου και να πολλούνται παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλωσορίζω το ότι αναμέναμε το να ε, έχουμε ελκυστήρες ε, με ψηλότερη ταχύτητα και επίσης έχουμε λύσει και το θέμα για το πώς θα έχουμε δύο κατηγορίες ελαφρών ε, οχημάτων, ένα για γεωργική χρήση και ένα για γενικότερη χρήση. Υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία μεταξύ των δύο εισηγητών και νομίζω η δική μου επιτροπή τα χειρίστηκε με ένα εξαιρετικό τρόπο το θέμα αυτό. Φυσικά δεν έχουμε τελειώσει ολοκληρώσει ακόμη, γιατί έχουμε και τις πτυχές του ελέγχου των κατεξουσιοδότηση πράξεων και θα δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι υπάρχει σε αυτές τις προτάσεις θα υλοποιηθεί ικανοποιητικά και θα καλύψει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Ευχαριστώ για ε, την ομάδα EFD. Μπάφτον για δύο λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σημαντικέ ανησυχίε σε σχέση με την επιλογή του άρθρου 18 που δεν μας ε, δίνει αποδείξεις ε, για ε, καταπολέμηση της νοφείας. Έχουμε την μελέτη αντικτύπου η οποία το αποδεικνύει αυτό. Μέσω του τριμερούς διαλόγου είχε τεθεί να γίνει μία εξαίρεση των οχημάτων ύπου 48 ύπων. Όμως αν εδώ δεν μιλάμε για πετήσεις αδειοδότησης και βασιζόμαστε εστιαζόμαστε μόνο σε στόχους περιβαλλοντικούς και ασφάλεια γιατί εξαιρούνται οι μηχανές 48 ε, ύπων ε, είναι κάπως κυκλικό το επιχείρημα. Καμία μελέτη αντικτύπου ε, για τις αγορές των εξαρτημάτων έχει γίνει. Αν μπορούν να απολυθούν στο μέλλον μόνο τα εξαρτήματα που έχουν τύχει έγκριση τύπου, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αιτιολογήσουν το κόστος της, του προϊόντος τους. Ε, ε, είχαμε μία, ένα έγγραφο το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο μέχρι σήμερα το πρωί το που παρουσιάζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα δεν ήταν στο δημόσιο ε, τομέα ούτε σε όλε τι γλώσσε αρκετά για να μπορέσουμε να το μελετήσουμε επαρκώ Η όλη διαδικασία είναι αμφιβόλου δημοκρατική νομιμότητα. Υπήρξε έλλειψη διαφάνεια, ε, γύρω από την νομοθεσία που προωθείται χωρίς ε, να υπάρξει αποτελεσματικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο πριν την αυριανή ψηφοφορία. Δόθηκαν από την Κομισιόν κάποιοι δημοσιονομικοί λόγοι, όμως ε, θα ήθελα να ζητήσω τουλάχιστον να αναβληθεί ψηφοφορία μέχρι μια ε, ορθή νομοθετική διαδικασία να ακολουθηθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο κύριος Σενίν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλοντας να ρυθμίσουμε τα πάντα, καθιστούμε τους κανονισμούς ανεπαρκής και ακατάλληλους. Μιλάμε για μοτοποδήλατα, για μοτοσυκλέτες, για δίκυκλα σαν να ανήκουν όλα στην ίδια κατηγορία. Ορισμένα από τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται ε, για άλλους λόγους και όχι για αυτούς που δημιουργήθηκαν. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε υποκατηγορίες. Ας πάρουμε τα τετράκυκλα. Όπως και οι μοτοσυκλέτες, τα τετράκυκλα έχουν γίνει μια πληγή τη σύγχρονης εποχής διότι χρησιμοποιούνται σε κατάλληλους χώρους χωρίς καθόλου ασφάλεια. Είναι λοιπόν επικίνδυνα τα οχήματα αυτά για τους πεζούς, για τα παιδιά και ε, παρόλο που δεν κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, ε, επειδή δεν κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά, δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 71% των θυμάτων τροχαίων που οφείλονται σε μινι quad ή μοτοσυκλέτες είναι παιδιά κάτω των 10 ετών. Αυτά τα οχήματα ε, προκαλούν συχνότατα ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση των οδηγών, στους κανόνες κυκλοφορίας με σκοπό να προστατεύσουμε τους οδηγούς που τηρούν τους κανόνες και τα, του, τα, το, το, το, τους κατοίκους, τους πολίτες που κινδυνεύουν να είναι θύματα καθημερινώς. Πρέπει λοιπόν να απαγορεύσουμε οποιαδήποτε εισαγωγή τέτοιων οχημάτων που δεν θα ανταποκρίνονται στους, στους, στους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα το... Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές που έχουν ζητήσει. Μίτσελ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές Βίμ Κάμπεν και Αντώνιο Πεντσέρη για τι εκθέσει Με αυτή την ευκαιρία και που είναι και ο επίτροπο εδώ θέλω να εκφράσω ανησυχίε σε σχέση με κάποιε πτυχέ προδιαγραφών ασφαλεία που προτείνει η Κομισιόν στο πακέτο ε, του Ιουλίου Φέτο. μόνο ε, τετράτροχα ε, υπόκειντο σε ε, δοκιμές ενώ τώρα έχουμε τρί και δίκυκλα ε, που θα υπόκεινται σε περιοδικές ε, εξετάσεις. αυτό που αναφέρθηκε στη μελέτη που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ότι μόνο 1% των ε, ατυχημάτων με τα ε, ε, δίκυκλα οφείλονται σε προβλήματα κατασκευής. Είναι σημαντικό όταν γίνεται αξιολόγηση προδιαγραφών ασφαλείας να συγκρίνουμε της, ε, την πρώτερη εμπειρία των χωρών ε, με σωστό τρόπο. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, είχαν το χαμηλότερο αριθμό ατυχημάτων, από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά δεν έχουν υποχρεωτικές δοκιμές ε, μοτοδικύκλων. Η Σουηδία είναι η μόνη σκανδιναβική χώρα όπου γίνονται περιοδικά ε, τεστ για να δουν αν μπορεί να κυκλοφορεί και αυτό άλλαξε το 2004 ε, και έγιναν κάθε δεύτερο χρόνο οι δοκιμές διότι είδαν ότι δεν χρειάζονται αυτά, αυτές οι δοκιμές τέτοια συχνότητα. Αυτή η απόφαση μέχρι τώρα από ό,τι μαθαίνω δεν επηρέασε αρνητικά τον αριθμό των ατυχημάτων στη Σουηδία από τα δίκυκλα. Επίσης για τους χρήστες των δικύκλων στην Ευρώπη το ε, κόστος ανέρχεται σε περίπου 1,2 δις για τη δοκιμή αυτή και αυτό ξεπερνά κατά πολύ ενδεχομένως τα ωφέλη. Ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε τον, την επίπτωση των δοκιμών στα τροχέα. Θα πρέπει πιστεύω να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα τη δύσκολη αυτή ε, ε, εποχή όπου το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο για τις οικογένειες. Επίσης τεχνικές ε, ε, προδιαγραφές για κάποια οχήματα θα πρέπει να στοχεύουν στην απλούστευση της νομοθεσίας και του διοικητικού φόρτου. Θα πρέπει να μπορέσουμε με εσωτερική εναρμόνιση να τα κάνουμε ασφαλέστερα τα δίκαικλα αυτά. Είναι σημαντικό να έχουμε εναρμονισμένες πολιτικές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μόνο όταν αυτές οι εναρμονισμένες πολιτικές έχουν θετικό και πραγματικό αντίκτυπο. Ευχαριστώ κύριε Τσικάου για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντικατεστούν τα εθνικά συστήματα έγκριση τύπου με μια διαδικασία ευρωπαϊκή έγκριση τύπου για να εγγυηθούμε την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου. Χρειάζεται ψηλό επίπεδο ασφάλεια, ασφάλεια στο χώρο εργασία αλλά και προστασία του περιβάλλοντο. Πρέπει λοιπόν να ενερμονίσουμε του τεχνικού κανόνε και τους περιβαλλοντικούς, ε, τα περιβαλλοντικά πρότυπα που αφορούν αυτά τα οχήματα αλλά και τα εξαρτήματα για την έγκριση τύπου και για τα γεωργικά και δασικά οχήματα αλλά και για τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα ο κανονισμός ε, και τα δίκυκλα, τρίκυκλα και τετράκυκλα εγγυάται μεγαλύτερη οδική ασφάλεια και βελτιώνεται και ο έλεγχος της αγοράς. Εμείς υπογραμμίζουμε ότι ο κανονισμός για την ε, έγκριση τύπου γεωργικών και δασικών χηματών ε, δεν θα πρέπει ουσιαστικά να διευκολύνει τη χρήση αυτών των χημάτων στους δημόσιους δρόμους θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ε, για να χρησιμοποιούνται αυτά τα οχήματα σε συγκεκριμένους δρόμους για να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό χρειάζεται πρόσβαση απερόριστη στις πληροφορίες σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση των οχημάτων και επίσης πρέπει να υπάρχει και ένας θεμητός ανταγωνισμός στην αγορά των επισκευών και πρέπει να παρέχονται και πληροφορίες για τη συντήρηση. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τεχνικές προδιαγραφές που να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ε, στις ιστοσελίδες ε, των κατασκευαστών. Εγώ θεωρώ θετικό το ότι η, η τροπολογία που προτείνεται από την Επιτροπή Μεταφορών όπου διαπιστώνεται ότι ένα όχημα ή ένα εξάρτημα όταν δεν σέβονται τις απαιτήσει αυτού του κανονισμού και δεν ε, λαμβάνει την έγκριση τύπου, τότε αυτό το προϊόν δεν θα τεθεί στην αγορά, ούτε θα επιτραπεί ε, να κυκλοφορήσει το όχημα και να ταξινομηθεί μέχρι ε, να είμαστε σίγουροι ότι σέβονται αυτά τα οχήματα τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ Μάνερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την εξαιρετική τους έκθεση. Για να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά είναι σημαντικό να έχουμε ε, μια εναρμονισμένη διαδικασία έγκρισης τύπου. Αυτό θα βοηθήσει τους κατασκευαστές ε, ελκυστήρων, γεωργικών ελκυστήρων, διότι η έγκριση τύπου Παραδείγματο χάρη, για τα γεωργικά και δασικά οχήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά ε, υπάρχει και το θέμα του κινδύνου. Μπορεί να συμβούν ατυχήματα και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα θέματα της ασφάλειας. Χρειαζόμαστε ασφαλή οχήματα διότι μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γι' αυτό χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα έγκρισης τύπου ώστε κάθε ε, αγρότης να μπορεί να, να χρησιμοποιεί μηχανήματα που είναι ασφαλή. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει και κάποια ευελιξία για τους εθνικούς κανονισμούς για τους μικρούς κατασκευαστές θα ήταν σκόπιμο να έχουν τη δυνατότητα ε, ε, ε, εθνικής έγκρισης τύπου, διότι αυτοί θα πουλάνε τα προϊόντα τους μόνο στο εσωτερικό των κρατών μελών. Τώρα, για τη μέγιστη ταχύτητα αυτών των οχημάτων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να ισχύσουν διεθνικές ρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρώση για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστήσω τους δύο και κυρίως τον το συνάδελφο Παντσέρη που έχει λειτουργήσει πολύ καλά ως διαμεσολευτή. Η συζήτηση αφορά δύο κανονισμούς με παρόμοια ζητήματα, την έγκριση τύπου γεωργικών δεσικών οχημάτων ε, και την έγκριση τύπου δικύκλων, τρικύκλων και τετράκυκλων. Η συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο μας οδήγησε ε, σε συμβιβεσμό και σε μια ομόφωνη πρακτικά ψηφοφορία. Ο στόχος είναι να πλουστευτεί η νομοθεσία, να έχουμε νέες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσει ε, και νέα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για γεωργικούς και δασικούς σκοπούς, ε, σκεφτήκαμε ότι καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός του, δεν χρειάζεται να έχουμε ε, υπερβολικές απαιτήσει τεχνικού και υπερβολοντικού χαρακτήρα. Βρήκαμε και μία συμφωνία για τα τετράκυκλα και τα χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες ε, για οχήματα αναψυχή και επαγγελματικά οχήματα και επίση έχουμε και τα δασικά οχήματα που πρέπει να προσαρμοστούν και να διαφορεθούν από τα προϊόντα τα οποία χρησιμεύουν για μεταφορά. Βρέθηκε ε, μία συμφωνία με του κατασκευαστέ ε, για την πρόσβαση σε πληροφορίε επισκευή και συντήρηση. ό,τι αφορά τι μοτοσυκλέτε, έχουμε περιβαλλοντικέ απαιτήσει, ε, όμω σημαίνει αυτό πρόσθετο άχθο για του κατασκευαστέ ενώ έχουμε ε, ουσιαστικά να αντιπροσωπεύουν το λιγότερο από 3% ε, των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δρόμο ε, για πολύ καιρό οι κατασκευές περίμεναν μαζί με τους χρήσεις πιο ξεκάθαρους και συγκεκριμένους και απλούς κανόνες που να μπορούν να εφαρμοστούν. Επομένως το αποτέλεσμα είναι θετικό. Ευχαριστώ. Γίνεις για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από το έργο του εισηγητού Βιμ Βαντεκάμπ. Ο Βιμ ο ίδιος είναι μοτοσυκλέτιστης και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έκθεση. Όπως ε, ως ε, σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΕ έλαβα πολλά email από μοτοσυκλετιστές πάνω στο θέμα. Και νομίζω ότι ο κύριος Βαντερ ε, βρήκε μια τη σωστή ισορροπία. Κυρία Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Κοινοβουλίου είναι να εξασφαλίζει την οδική ασφάλεια. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα, τη ρύθμιση για τα ABS και CBS συστήματα και για το γεγονός ότι υποχρεωτικά θα διασφαλίζεται ότι τα φώτα πορεία την ημέρα θα είναι σωστά τοποθετημένα. Ξέρουμε ότι οι μοτοσυκλετιστές έχουν οχταπλάσιο κίνδυνο να εμπλακούν σε ατύχημα σε σχέση με τους οδηγούς άλλων οχημάτων. Αυτό είναι αναντήρητο. Ελπίζω ότι οι μοτοσυκλετιστές θα μπορέσουν να καταλάβουν το νόημα αυτού του κανονισμού και γιατί έχει τόση σημασία. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ε, ε, καλό τριμερή διάλογο μεταξύ Κομισιών Συμβουλίου και του κυρίου Βαντεκάμπ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παρόλο που καμιά φορά ήταν βραδύς αυτός ο διάλογος, ε, τελικά έχουμε τις κατάλληλες και ακριβείς ρυθμίσεις. Και ως Ευρωπαίοι πρέπει όλοι να εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι θα μειωθούν ε, οι θάνατοι στους δρόμους μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την άλλη έκθεση του κυρίου Παντσέρη, τους ελκυστήρες ε, και τους, τα δασικά οχήματα, είμαι αρκετά ικανοποιημένος ότι ο εισηγητής επέτυχε καλή ισορροπία για να αποφύγει την υπερβολική γραφειοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση αυτή είναι αποτελεσματική σε σχέση με το περιβάλλον, την εσωτερική αγορά, αλλά και την, ε, το διασυνοριακό εμπόριο ελκυστήρων. Πρόεδρε, ελπίζω πραγματικά ότι έτσι θα, έχουμε, θα, θα δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική αγορά για τους ελκυστήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα έχουμε το ΚΑΤΣΔΙΑΙ. Μπασέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων για τα οποία είναι υπεύθυνα οι μοτοσυκλετιστές είναι υπερβολικά υψηλός και πρέπει να μειωθεί. Αυτοί οι οδηγοί διατρέχουν ε, πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτων. Γι' αυτό χρειάζεται μια πλούστευση του νομικού πλαισίου και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα περιβάλλοντος, ασφάλειας και ελέγχου της αγοράς. Ταυτόχρονα πρέπει να μην ξεχνάμε τη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ε, αστική κινητικότητα πιο πράσινη και πιο αποτελεσματική ε, είναι, είναι πολύ σημαντικές οι προτάσεις διότι θα μας εξασφαλίσουν μεγαλύτερη παρακολούθηση της ε, εσωτερικής αγοράς και για να γίνει αυτό χρειάζονται δεσμευτικά κριτήρια. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ε, ελπίζω ότι θα έχουμε για τα μοτοποδήλατα ένα πιο σαφές πλαίσιο ώστε να προστατεύονται οι οδηγοί οι οποίοι ε, κυκλοφορούν στους δρόμους. Υπάρχουν και πλεονεκτήματα, πρέπει να εξηγήσουμε τα πλεονεκτήματα των αποφάσεών μας στους ψηφοφόρους μας. Πρέπει να ε, έχουμε σαφή στοιχεία για την ασφάλεια των διαφόρων μερών ενός οχήματος ή ενός μοτοποδήλατου. Έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλεγχος και αξιολόγηση επιπτώσεων. Διάβασα αυτή την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να επειδή δεν με ικανοποίησε, δεν με ικανοποίησε η απάντηση της Επιτροπής, θα τη ζητήσω για μια ακόμη φορά να μου υποβάλει όλα τα στοιχεία ώστε να ενημερώσω σχετικά τους ψηφοφόρους μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τσουρνέσκι, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Απόψε είναι η Ιταλική βραδιά. Η πρόεδρος ε, ε, από την Ιταλία, ο Επίτροπος Ιταλός και συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και εγώ λαμβάνω τον λόγο ως μέλος της Επιτροπής Μεταφορών. Πιστεύω ότι η απόψινή μας συζήτηση έχει τεράστια σημασία. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να ρυθμίζουμε τα πάντα με τους νόμους. Εγώ είμαι κατά της υπερβολικής ρύθμισης. Όμως αυτοί οι κανονισμοί είναι απαραίτητοι και χρειάζονται λόγω του υπερβολικά μεγάλου αριθμού των θανάτων και στην Πολωνία, ε, στους δρόμους μας. Ε, έχουμε συνάδελφο που κόντεψε να σκοτωθεί σε ε, ατύχημα με μοτοσυκλέτα. Κρίμα που δεν είναι παρόν γιατί θα προσυπέγραφε αυτά που λέω. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εγκριθεί αυτή η νομοθεσία. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ. Η απλούστευση έγκριση τύπου για τα μικρά οχήματα, τα αματοποδήλατα, δίκυκλα, τρίκυκλα είναι καλά νέα για τους ε, χρήστες, δεδομένου ότι δεν θα καταστήσει πιο δύσκολη τη ζωή τους παρόλα αυτά, οι κατασκευαστές και οι πολιτές, οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες προκλήσεις, γιατί τα υποχρεωτικά συστήματα ε, πέδηση αντιεμπλοκή ε, σίγουρα θα σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλότερο κόστος ε, και θα αναγκαστούν οι κατασκευαστές να εξυγχρονίσουν περισσότερο την παραγωγή τους και έτσι τα προϊόντα θα είναι ε, πιο ακριβά λόγω των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Όμως ε, θα βελτιώσουμε ε, την ασφάλεια και αυτό ουσιαστικά θα αντικατοπτρίσει, θα ε, έρθει να αντισταθμίσει την υψηλότερη τιμή χάρη στην νομοθεσία. Ελπίσουμε όμως ότι θα το καταλάβουν το ίδιο και οι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Αν δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Ταγιάννη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία σε έθεσε ένα πρόβλημα ότι αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνεται σε ένα ειδικό γραφείο, όμως στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί έχουμε πολύ σημαντικά πολιτικά αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν εγκρίνοντας αυτά τα δύο νομοθετήματα και πρόκειται κυρίως ε, για κανόνες που θα συμβάλλουν στο να έχουμε περισσότερη οδική ασφάλεια. Θα προστατεύουμε λοιπόν ε, τους πολίτες μας. Πρόκειται για κανόνες που απλουστεύουν ε, την προηγούμενη νομοθεσία και αυτή είναι μια ακόμη επιλογή που επίσης ευνοεί τους πολίτες και επίσης πρόκειται για κανόνες που συμβάλλουν στην ε, καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος ε, και βοηθούν και, και τις επιχειρήσεις μας, είτε είναι μικρές είτε μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω κυρίως από τη σκοπιά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όπως ε, υπενθυμίστηκε από κάποιους κυρίως βουλευτές ε, ότι ε, πρέπει να ε, δούμε το πολιτικό αποτέλεσμα στην έγκριση τύπου και στις δύο ομάδες είχαμε μία ταχεία διαδικασία από τη σκοπιά της δεσμευσής της νομοθετικής ε, έχουμε πετύχει καλά αποτελέσματα. Πρόκειται για ουσιαστικούς παράγοντες για να έχουμε ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα και που θα εγγυηθεί στο να κυκλοφορήσουν στην αγορά οικολογικά οχήματα προσφέροντας ε, και επιπλέον ωφέλη στους ε, κυρία δεν είναι εδώ, αλλά θα αναφερθώ στο θέμα που έθεσε σε σχέση με την ε, παραποίηση. Ε, εγώ έχω λάβει κάποια στοιχεία από την Ιταλική Δημοκρατία ε, σε σχέση με προσπάθειες καταπολέμησης παραποίησης και θέλω να επαναλάβω ότι όχι μόνο στον κλάδο των παιχνιδιών ή στον τομέα των υποβημάτων αλλά και στα αυτοκίνητα υπάρχουν τέτοιε παραπείσεις και θέλω να υπενθυμίσω ότι το κείμενο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για το ΚΑΡΣ 2020 με δεσμεύει στο να προχωρήσω προς την εποπτεία ε, της παραποίησης της εσωτερικής αγοράς ε, με την ίδια αποφασιστικότητα και αυτό θα πράξουμε και για τους δύο τομείς ε, οχημάτων, για τις κατηγορίες οχημάτων που συζητούμε σήμερα, με στόχο να βελτιώσουμε τις νομοθετικές διατάξεις που θα απλουστεύουν ε, την κατασκευή και ε, θα βοηθούν την αλυσίδα προμήθειας. Επίσης θα υπάρξει ενοποίηση των συστημάτων έγκρισης τύπου των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αστυνομία, επομένως ε, θα το αναθέσουμε όλα αυτά στα κράτη-μπέλη προκειμένου να εποπτεύουν για την καταπολέμηση της παραποίησης. Μια άλλη δέσμευση είναι υπάρξει ένα φόρουμ για να συντονίσουμε τις δράσεις εποπτείας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το σημείο ενίσχυση των απαιτήσεων ε, στον τομέα του ανταγωνισμού και παροχή τεχνικών ε, τεχνικών που να βελτιώνουν τα συστήματα έγκρισης τύπους. Επίσης θα στείλουμε όλες τις πληροφορίες που ζητήθηκαν ε, προκειμένου να ενημερώσετε και τους ψηφοφόρους σας. Ε, λυπάμαι που βγήκε από την αίθουσα. Ε, θα έρθουμε όμως σε επαφή μαζί του για να του δώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ νέου τους δύο συγητές. Δεν ε, μπορώ να δωρήσω μια μοτοσυκλέτα στον ε, κύριο Βαντεκάμπ ή έναν ελκυστήρα στον ε, κύριο Παντσέρη, αλλά πιστεύω ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα δικυκλά και τις μοτοσυκλέτες θα χαρούν πάρα πολύ για το έργο που υλοποιήθηκε για να γίνει, ουσιαστικά να γίνουν τέτοιες βελτιώσεις σε αυτά τα οχήματα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή Βάντεν Κάμπ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τις απαντήσεις που μας έδωσε και τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν όλοι γυρίσει, αποχωρήσει για τα κομπλιμέντα και την υποστήριξη που μου έδωσαν για αρκετό καιρό. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή αυτά που μας είπε ο Επίτροπος. Μας είπε ότι θα φροντίσει να προωθηθεί το θέμα και, σε ό,τι, και δεν θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνος για τις ε, εκτελεστικές πράξεις και τις πράξεις κατεξοδότηση ώστε να μπορέσει η βιομηχανία να εφαρμόσει τους νέους κανόνες και τις νέες ρυθμίσει. Δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην έρευνα σχετικά με το σύστημα BS για τα μικρά σκούτερ ή το, τι θα γίνει με το πρότυπο ε, Euro 5 μέχρι το 2015 αλλά ελπίζω ότι θα το λάβει υπόψη και θα μας απαντήσει σχετικά. Και θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε αυτή τη φάση της συζήτησης. Η ανακοίνωση για το νέο κανονισμό θα είναι σαφής, διότι ε, μιλάμε για μια ουσιαστική σημαντική απλούστευση. Θέλουμε η ενημέρωση για τη συντήρηση και τις επισκευές να είναι προσιτή σε όλους και είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό να προσδιοριστεί με σαφήνεια. Ε, στον Άγγλο συνάδελφο Εύτον ε, θα ήθελα να πω ότι αν είχε συμμετάσχει νωρίτερα, νωρίτερα στη συζήτηση θα μπορούσε να έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα. Τον βλέπω για πρώτη φορά απόψε. Κρίμας. Ακόμα κάτι είναι γεγονός ότι αγόρασα ε, μια νέα μοτοσικλέτα BMW είναι, αυτό είναι πολύ καλό για την ε, ε, ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία σημαίνει ότι θα έχουμε μία ιαπωνική μοτοσυκλέτα λιγότερη. Ο κύριος Παντσέρη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Ταγιάννη, για όσα είπε. Δεν θα ήξερα τι να το κάνω το τρακτέρ, το ελκυστήριο έτσι λοιπόν καλύτερα να μείνει και που είναι. Δεν ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε κάτι παραπάνω. Είδαμε από τη συζήτηση πώ συνένεση υπάρχει γύρω από τα ζητήματα αυτά για την έγκριση γεωργικών και δασικών εχμέτων και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί εργαστήκαμε για να υπάρξει μια τέτοια συνένωση και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε. Ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στι 12 το μεσημέρι. Επόμενη συνεδρίαση θα γίνει αύριο, 3η 20 Νοεμβρίου, από τις 8.30, ε, από τις 12.30, από τις 3.